του δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 και δίνω το λόγο στην Ιζαμπέλ Τωμά. Μια στιγμή κυρία Τόμα. Περιμένετε μια στιγμή να αποχωρήσουν οι συνάδελφοι. Σας παρακαλώ να αποχωρήσετε ηρέμος, ησύχος και σιωπηλός και το ταχύτερο δυνατό λέει ο πρόεδρος. Κυρία Φανμπρέμπτ. Mm. Κυρία Φανμπρέμπτ. Κυρία Λούνατσεκ, παρακαλώ, ή να καθίσετε ή να φύγετε. Πάρτε και την κυρία Βαν Μπρέμπτ μαζί σας αν μπορείτε. So. Ο Τωμά, πείτε. Κύριε Τωμά, έχετε το λόγο. Ε, Madame la Commissaire, chers collègues, nous sommes aujourd'hui face à... Κυρία Επίτροπε, κυρίε και κύριοι, το θέμα που μας απασχολεί είναι αρκετά τεχνικό αλλά έχει και πολιτική σημασία στα ισχύοντα προγράμματά μας. Όλα τα διαχειριστικά ταμεία 14-20 αφορούνται. Στην 31 Δεκεμβρίου του 2014 πάνω από 300 ε, προγράμματα δεν είχαν ακόμη εγκριθεί και επομένως ε, θα τους εφαρμοζόταν η αναβολή ή μεταφορά κονδυλίων. Όλα τα κράτη-μέλη ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα. 21 δισεκατομμύρια ευρώ θα χαθούν χωρίς την αναθεώρηση. Για μερικά κράτη αυτό είναι πολύ ουσιώδες, οι δεσμεύσεις δηλαδή, οι προβλέψεις. Παραδείγματα, για την Τσεχία 99% των ποσών θα χάνονταν για τη Ρουμανία 80% για την Ισπανία πάνω από 60% και πάνω από 50% για το Ηνωμένο Βασίλειο ευτυχώς το άρθρο 19 του Πολδίπ επιτρέπει τροποποιήσεις μέχρι την 1η Μαΐου μέχρι την 1η Μαγιά για να αλλάξει η κατανομή των κονδυλίων εφόσον δεν υπάρξει προσαρμογή για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν είμαι υπέρ της αναθεώρησης που θα ψηφίσουμε. Λόγω όμως των περιφερειακών επιπτώσεων που θα έχουν όλα αυτά σε όλες τις χώρες, η αναθεώρηση αυτή προστίθεται σε δυσλειτουργίες ανησυχητικές. Πρώτον, τίθεται ακόμα μια φορά το θέμα της ε, ειλικρίνειας των δημοσιονομικών μας διαδικασιών γιατί το ξέραμε ότι θα είχαμε καθυστερήσει. Δεύτερον, επειδή είναι χρόνιο το έλλειμμα, μια τέτοια καθυστέρηση των διαρθρωτικών ταμείων που συνδέεται για, με την κύρωση των λειτουργικών προγραμμάτων είναι απαράδεκτη. Τρίτον, αυτή η καθυστέρηση της εφαρμογής θα έχει επίπτωση και στις πληρωμές διότι οι δεσμεύσεις μπορούν να καθυστερήσουν ένα χρόνο αλλά οι πληρωμές όχι γιατί έτσι αυξάνεται ακόμα περισσότερο η πίεση και μάλιστα σε την περίοδο που λύγει το δημοσιονομικό πλαίσιο. Όλη αυτή η χιονοστιβάδα λοιπόν αμφισβητεί, θέτει ένα αμφιβόλο την αξιοπιστία της Ένωσης και θα θέλω, θέλω να το καταλάβετε ότι η αναθεώρηση δεν χειροτερεύει το θέμα των ελλημάτων αλλά μπορεί να αυξήσει τα προβλήματα στο τέλος της περίοδου και χαιρετίζω εδώ τη δήλωση της Κομισιόν ότι θα χρησιμοποιήσει ό,τι ευελιξία διαθέτει για να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις της αναθεώρησης. Παρ' όλα αυτά κυρία Επίτροπε φοβάμαι ότι η ευελιξία αυτή δεν θα αρκέσει. Το Κοινοβούλιο είχε ήδη εκφράσει τους φόβους και τις ανησυχίες του από το 2013 και για πρώτη φορά σημειώνεται τέτοια μείωση και αυτό δείχνει ότι δεν έχουμε προσαρμοστεί. Χρειάζονται λοιπόν ορισμένες δημοσιονομικές προσαρμογές που όλες μαζί αποτελούν την αναγκαιότητα, δείχνουν την αναγκαιότητα της αναθεώρησης και πολιτικής και δημοσιονομικής. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατικών Επενδύσεων και το απόθεμα ευελιξίας θα επηρεαστούν και αυτά. Όλοι εδώ γνωρίζετε ότι δεν είναι ειλικρινές το Συμβούλιο ως προς τον προϋπολογισμό και ότι ο ετήσιος χαρακτήρας του έχει τεθεί ένα στην πράξη. Με την αναθεώρηση λοιπόν αυτή έχουμε την μια ιστορική ευκαιρία, όχι αυτή την τεχνική αναθεώρηση, την πολιτική αναθεώρηση που μας περιμένει. Αυτή η ευκαιρία ή αυτό το καθήκον στηρίζεται σε τρία στοιχεία. Πρώτον, οι εκλογές έδωσαν ένα μήνυμα στους εκλογείς ότι αμφισβητούν ή και απορρίπτουν την Ένωση. Δεύτερον, η οικονομική κρίση απαιτεί μια αντιμετώπιση με τον δέοντα τρόπο και αυτό το βλέπουμε από τις συζητήσεις για το ΕΦΣΥ Τέλος, το δημοκρατικό έλλειμμα. Ποιες είναι οι πολιτικές ευθύνες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε ως νομοθέτες. Έχουμε ποτέ ξαναδεί κοινοβούλιο να ψηφίζει πάνες χωρίς να αναρωτιέται για τα αντίστοιχα έσοδα. Εδώ είναι ο κόσμος ανάποδα. πρέπει να διασφαλίσουμε και τα έσοδα χωρίς πρόσθετους φόρους. Αυτή τη στιγμή οι φορές είναι το 75% του προϋπολογισμού και αυτό εκτρέφει τις ιδέες εκείνων που ζητούν την λεγόμενη δίκαια ανταπόδοση. Η κρίση των πληρωμών καθιστά τον ε, ενωσιακό προϋπολογισμό απλό βοήθημα για τους εθνικούς και αυτό δείχνει, δίνει πολύ άσκημα σημάδια στους λαούς της Ευρώπης. Έχω ένα λεπτό ακόμα αλλά δεν θα το χρησιμοποιήσω κύριε Πρόεδρε για τα συμπεράσματα. Πρέπει κυρία Επίτροπε να πούμε ότι πρέπει να επανέλθουμε σε αληθινούς ιδίους πόρους με το αντίστοιχο κοινωνικό πρόγραμμα. Κυρία Πρόεδρε, ζητώ μια πραγματική αναθεώρηση μετά τις εκλογές και αυτό οφείλεται στο ότι συμμερίζομαι το αίσθημα ακριβώ της Κομισιόν ότι βρισκόμαστε σε καμπή της ευρωπαϊκής οικοδόμησης και βλέποντας μπροστά μας την αύξηση των λαϊκισμών δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να αποτύχει ως προς αυτό. Χρειάζεται μια πολιτική αναθεώρηση του προϋπολογισμού για το 2016 και μπορείτε να υπολογίζετε στη στήριξη όλων των δημοκρατών εδώ μέσα. Φερνάντες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να χαιρετήσω την παρουσία της κυρίας Επιτρόπου. Θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όλους τους συναδέρφους που έχουν βοηθήσει στο έργο αυτό. Έχουμε μπροστά μας μια εξόχως τεχνική πρόταση, η οποία όμως ενεκρίθη ομόφωνα <clears throat> στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Είναι μια πρόταση για την οποία θα πρέπει να εκφράσουμε και κάποιες πολιτικές σκέψεις για το μέλλον. Οι καθυστερήσει στο δημοσιονομικό πλαίσιο στην έγκρισή του οδήγησε σε καθυστέρηση στα λειτουργικά προγράμματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική συνοχής. Οι πόροι της ε, ε πολιτικής συνοχής, πόροι, πόρη, πόρη αγροτικής ανάπτυξης, το Ταμείο Αλλιευτικής Ανάπτυξης Αυτά ήταν τα κονδύλια τα οποία επλήγησαν περισσότερο και η πολιτική συνοχή επίσης, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για όλους μας. Είναι λοιπόν σημαντικό, είναι κατεπήγον όλα αυτά τα λειτουργικά προγράμματα σε περιφερειακό επίπεδο, ιδίως τα λειτουργικά προγράμματα τα οποία αφορούν την πολιτική συνοχής, το Ταμείο Συνοχής και το Κοινωνικό Ταμείο να μπορέσουν να εφαρμοστούν με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Σας υπενθυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάνω από 200 περιφέρειες αλλά ένα μεγάλο μέρος από αυτές βρίσκεται κάτω από το 75% του ε, μέσου όρου του ΑΕΠ κατά κεφαλήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περίπου μία σε κάθε τέσσερις περιοχές είναι μία με, με χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης περιοχή της Ευρώπης. Είναι απαραίτητο λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ασυμμετρίες και να έχουμε μια νέα μορφή προσέγγισης και ένα νέο τρόπο δράσης των ταμείων αυτών μέσα σε ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο για να μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερο έναυσμα στην οικονομική ανάπτυξη, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί μια προτεραιότητα στην ευφυή στις ευφυείς μορφές ανάπτυξης. Σήμερα η πολιτική συνοχή σημαίνει χαινοτομία, σημαίνει νέες ενέργειες και προσπάθειες. Δεν πρέπει να χαθούν λοιπόν οι πόροι οι οποίοι οδηγούν σε προσθέμενη αξία για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε εδώ για μια μεταφορά πιστώσεων που δεν είναι ουσιαστικά ε, πληρωμές, είναι απλώς μεταφορές δεσμεύσεων υποχρεώσεων. 21,1 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν το 2015 και το 2016. Είναι απαραίτητο λοιπόν τα προγράμματα αυτά τα λειτουργικά τα οποία ανέφερα αλλά και τα προγράμματα και το Ταμείο για το Άσυλο και την ε, Μετανάστευση, για την Ενσωμάτωση και για την Εσωτερική Ασφάλεια να βρεθούν σε λειτουργία το ταχύτερο δυνατό. Αυτή λοιπόν η τροποποίηση του δημοσιονομικού πλαισίου, αυτή η μεταφορά πιστώσεων θα μας επιτρέψει σε αυτά τα 300 προγράμματα να μην παραμείνουν καθυλωμένα λόγω των καθυστερήσεων που έχουν ήδη επισυμβεί. Είναι απαραίτητο επίσης να υπογραμμίσω <clears throat> ότι το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο απαιτεί ευκαμψία, απαιτεί μία αναθεώρηση, μια τροποποίηση που να λάβει υπόψη της ε, υποστήριξης της ανάκαμψης οικονομικής, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και να υπάρξει και υποστήριξη σε νέα σχέδια όπως το σχέδιο Juncker. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να μας οδηγήσουν σε μια εξέταση ποιον ποιες γραμμές του προϋπολογισμού θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πιο επωφελώς για το σχέδιο Juncker. Αυτή λοιπόν η αναθεώρηση είναι μια μεγάλη ευκαιρία του πολιετούς ε, προγράμματος. Ελπίζω ότι και στην Ολομέλεια θα γίνει δεκτή αυτή η αναθεώρηση με την ίδια συνένεση και ομοφωνία όπως στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα σας είναι ευγνώμονες εάν το πράξετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Φερνάντες λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα. Η Ιωσταλίνα Γεωργίευα, την πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και επίση να ευχαριστήσω θερμότατα την εισηγήτρια, την κυρία Τομά. Αλλά Ευχαριστώ ευχαριστήσω και τον κύριο Φερνάντε, διότι ε, ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρο αυτό το οποίο εξήγησαν για τη σημασία ε, αυτή τη προτινωμένη ε, αλλαγή στον πολιτισμό όσον αφορά την Ευρώπη και για το πόσο επήγει η σχετική απόφαση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τα κρατημέλη κατέβαλαν πάσα δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε να εγκρίνουν όσο γίνεται περισσότερα προγράμματα το 2013. Και αυτό είπαμε πριν πρέπει να συνοδεύεται από υψηλή ε, ποιότητα όσον αφορά την ε, απορρόφηση και την χρησιμοποίηση των κονδυλίων. Και προσπαθούμε να κάνουμε κάτι και πριν ε, επιληφθεί το θέμα στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο γιατί θα πρέπει να σας πω επίση ότι προσπαθήσαμε για το, συγγνώμη, για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο πριν ισχύσει το ε, δημοσιονομικό πλαίσιο μπορούσαμε κάτι να κάνουμε και αυτό το κάναμε και για το επόμενο αλλά και για το προηγούμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Έχουμε επίσης και τον ε, κανονισμό του Συμβουλίου για ε, αυτό το δημοσιονομικό πλαίσιο ε, για την περίοδο 2014-2020 επίσης έχουμε και κάποιες καθυστερήσεις όσον αφορά την νομοθέτηση των σχετικών πράξεων αλλά αυτό είχε αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά διάφορα προγράμματα, διότι έχουμε το 47% των προγραμμάτων τα οποία επλήγησαν, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν εγκριθεί και να τρέχουν το 2014. Όπως ήδη αναφέραμε, πρόκειται για 21,1 δις ευρώ. Και επομένως χάθηκαν 6 μήνες λόγω αυτής της καθυστέρησης και αυτό το οποίο θέλουμε να προτείνουμε αυτή την τεχνική προσαρμογή να υπάρξει περισσότερη ευελιξία για να παραταθεί η σχετική περίοδος και έτσι να μας δοθεί το περιθώριο ακριβώς όπως λέει στο 19 του κανονισμού του Συμβουλίου για την αναθεώρηση του ε, κανονισμού αυτού πριν από τον Μάιο του 2015. Θέλω τώρα να σας αναφέρω τα εξής τρία. Πρώτα πρώτα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάρα πολύ σκληρά για να επιταχυνθεί η έγκριση για να έχουμε περίπου 16 δις για το 2015 και τα υπόλοιπα όπως προτάθηκε ε, και όπως εγκρίθηκε να μεταφερθούν το 2016. Κατά δεύτερο λόγο επίσης ε, θεωρούμε πάρα πολύ θετικό το ότι η Επιτροπή των Προεδρικών του Κοινοβουλίου πήρε το θέμα πάρα πολύ ζεστά και δούλεψε γρήγορα για να κατέβει η σχετική πρόταση εδώ στην Ολομέλεια. Οπότε και εγώ όπως και οι συγκητέ, ελπίζουμε ε, η ψηφοφορία να είναι θετική επίσης και ο κ. και η κυρία Τομά ε, μίλησαν για το πόσο χρειάζεται να ε, χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευελιξία που μας προσφέρεται. Αυτό που, για το οποίο έχει παλέψει το Κοινοβούλιο να γίνει αυτή η προσαρμογή του πολιετούς πλαισίου κατά τις επόμενες χρήσεις. Οπότε είπαμε, όπως είπε και η Επιτροπή αυτή, να γίνει μια μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση, οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ στα σοβαρά θα εργαστεί σε μια πρόταση που θα την ε, υποβάλει όταν έρθει η ώρα. Οπότε, όπως είπαμε, όλα αυτά ήταν πολύ σημαντικά και είπαμε τα κάνουμε όλα όσο γίνεται με πιο επίγοντα ρυθμό για την οικονομία, για την απασχόληση, για τη βελτίωση της ζωής των Ευρωπαίων οπότε και εμείς ε, ε, ε, θα στείλουμε το λόγο μας ότι πρόκειται το συντομότερο δυνατόν να εγκρίνουμε αυτή την αναθεώρηση και να εξασφαλίσουμε το ότι θα ρεύσει το, χρήμα προς τα προγράμματα που θα δώσουν ευκαιρίες για απασχόληση και ανάπτυξη στην Ευρώπη. Ο Πρόεδρος. ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση αυτή, κυρία Αντιπρόεδρε. Από την Περιφερειακή Επιτροπή τώρα ο κύριος Μποστινάρου. Κυρία Επίτροπε, επιτρέψτε μου να μιλήσω στην Ρουμανική. Από την αναθεώρηση του Πολδίπ τίθεται ε, η αναθεώρηση του πολυδίπου είναι προϋπόθεση για να μην χαθούν κονδύλια του 2014 για μια ολόκληρη σειρά προγραμμάτων που δεν μπόρεσαν να απορροφηθούν λόγω καθυστερήσεων. Είμαι πεπισμένος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει υπέρ της αναθεώρησης. Η πολιτική συνοχή είναι από εκείνες που έχουν πληγεί πιο πολύ από τις καθυστερήσεις και που αφορούν και τα υψηλότερα ποσά επειδή πρόκειται για πολιτική επενδύσεων που είναι η πιο αποτελεσματική μέχρι στιγμή στην Ένωση πρέπει οπωσδήποτε να γίνει η αναθεώρηση. Να μην χάσουμε άλλο χρόνο ώστε η εφαρμογή των προγραμμάτων να αρχίσει όσο δυνατόν συντομότερο προλογισμό του 2015 θα πρέπει να τροποποιηθεί επίσης και ζητώ από την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να καταλήξουν όσο το δυνατόν συντομότερα τα προγράμματα προσαρμογής για να σταματήσουν οι καθυστερήσεις. Και ζητώ από την Κομισιόν να μας ε, βεβαιώσει ότι δεν θα συνεχίσουν να συσσωρεύονται οι καθυστερήσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαστε ήδη στα μέσα Απριλίου και η κατάσταση είναι ανησυχητική και μας αναγκάζει να αναθεωρήσουμε γραφειοκρατικές και άχρηστες διαδικασίες που, που δημιουργούν τις καθυστερήσεις. Και μάλιστα να λύσουμε αυτό το πρόβλημα κατά προτεραιότητα ώστε να μην υπάρξει ανάλογο και στο μέλλον. Έτσι θα πρέπει να αναθεωρηθεί και το χρονοδιάγραμμα. να απομένουσες πληρωμές πρέπει και αυτές να μπουν μέσα στο πλαίσιο της μεσοπρόθεσμης αναθεώρησης. Προβλέπεται η μεταφορά 21 δισεκατομμυρίων από το 2014 και θα ήθελα να προσέξουμε ότι έτσι αναγκάζουμε τα κράτη-μέλη να απορροφήσουν πολύ περισσότερα κονδύλια με κίνδυνο να μην αναλυφθούν περαιτέρω δεσμεύσεις. Από την άλλη πρέπει να καταλάβουμε ότι το μεγάλο ύψος των καθυστερήσεων και των καθυστερουμένων πληρωμών για τα διαρθρωτικά ταμεία και τις επενδύσεις δημιουργούν με τη σειρά τους ακόμα περισσότερη ανάγκη άμεσων πληρωμών. Για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει η Κομισιόν να διασφαλίσει ότι τα εκρεμή ποσά θα απορροφηθούν από το 15 μέχρι και το 17 Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες στην εφαρμογή των επενδύσεων και στις περιφέρειες και για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Πρέπει να αποδειχθεί, επιδειχθεί πνεύμα συνεργασίας ώστε να μπορέσουν να εφαρμοστούν και τα καθυστερούμενα προγράμματα με την αναγκαία χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκριτιθάμπολ μάλλον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ακριβώ όπως αναφέρθηκε τώρα συζητούμε αυτή την τροποποίηση του δημοσίου πλαισίου. Πάρα πολύ σημαντικό τόσο ώστε να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε αυτά τα 21 δι ευρώ. Αυτά τα οποία για διαφορετικού λόγους δεν μπορέσαμε να χρησιμοποιήσουμε το 2014 να μεταφερθούν το 2015. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούν θα πρέπει να γίνει σύντομη έγκριση και το σημαντικό είναι να αρχίσουν να τρέχουν αυτά τα προγράμματα. Αυτό το οποίο τώρα θέλουμε είναι να σας πω το τι θα γίνει με τις πληρωμές. Ε, όχι μόνο με αυτή την αλλαγή στο δημόσιο πλαίσιο, αλλά για το τι γίνεται όσον αφορά τη μεταφορά των πιστώσεων γιατί αυτή η συζήτηση την οποία κάνουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφορά αυτές τις ε, πληρωμές και αυτό είναι για τις ε, πληρωμές που δεν έχουν γίνει. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το δημοσιονομικό πλαίσιο, πώς θα σταθεροποιηθεί η ε, πώς θα, γίνει η πληρωμή γιατί είπαμε ότι με αυτή την τροποποίηση ε, και με την καθυστέρηση της, της ε, λειτουργίας των προγραμμάτων έχουμε αυτή την υπέρβαση αλλά αυτό το οποίο θέλαμε να κάνουμε είναι το 2014 να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα οποία ε, έπρεπε να χρησιμοποιούν στο τέλος της θητείας αλλά θα πρέπει να γίνει καλύτερος προγραμματισμός οπότε γι' αυτό και αυτή η αναθεώρηση που είπαμε είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το λάβει υπόψη η Ευρωπαϊκή Οτρία και να υπάρχουν αρκετά κονδύλια ούτως ώστε να μην ξαναπέσουμε στην ίδια θλιβερή κατάσταση όπως συνέβη προκειμένου. Κούσμιουκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, εδώ και 1,5 έτος έχουν εγκριθεί οι δημοσιονομικές προοπτικές 2014-2020. Ε, Πολλά λειτουργικά προγράμματα λοιπόν σε τομείς διαδοτικούς και στη γεωργία έχουν προετοιμαστεί από τα κράτη-μέλη και έχουν υποβληθεί στην Κομισιόν. Υπάρχει όμως μια μεγάλη καθυστέρηση σε 300 και πλέον προγράμματα αυτού του είδους. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει ένας αναπρογραμματισμός για τις δημοσιονομικές προοπτικές στα επόμενα χρόνια. Πρέπει λοιπόν να ετοιμάσουμε διορθωτικούς προϋπολογισμούς υπαριθμών 2 για το 2015 που θα επιτρέψει να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα 21,1 εκατομμύρια ευρώ πιστώσεων υποχρεώσεων από το 2014 και να τα μεταφέρουμε το 2015. Αυτό θα επιτρέψει να καταβληθούν οι πληρωμές το 2015 και 2016. Θα ήθελα να πω σχετικά ότι αυτή τη στιγμή είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε στην ταχύτερη δυνατή υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών και να χρησιμοποιηθεί πλήρω το δημοσιονομικό πλαίσιο. Η μεταρρύθμιση αυτή να γίνει το 2016 για να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Ο κύριος Ντεπρέ. Κυρία Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ τους δύο συγητές, την κυρία Τομά και τον ε, κύριο Φερνάντης ιδίως τον τελευταίο, γιατί αυτός είναι ο οποίος έχει επομιστεί την γενική ευθύνη για, τους, ε, ε, για τις εκθέσεις προϋπολογισμού που αφορούν το ΕΛΚ. Υπάρχει το άρθρο 19 σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό κανονισμό. Πρόκειται για 21 εκατομμύρια ε, πιστώσεων υποχρεώσεων, τα οποία θα είχαν ακυρωθεί χωρίς αυτή τη δυνατότητα μεταφοράς και δεν θα ήταν ε, χρησιμοποιήσιμα για την επιμερισμένη διαχείριση. Πολύ σωστά. Αλλά να, κάνω και μία, να εκφράσω και μία άποψη. Εγώ βρίσκω πραγματικά εκπληκτική αυτή τη συνήθεια που έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να κάνουμε τέτοιου είδους τροποποιήσεις όχι μονάχα σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, αλλά και σε ό,τι αφορά τις νομικές βάσεις και την τροποποίηση των διαδικασιών. Αυτό σημαίνει πάλι κάποια διαδικασία μαθητείας για τις δημόσιες αρχές για να ε, λειτουργήσουν. Κάθε 7 χρόνια τα κάνουμε όλα τα μπουλαράζα, τα κάνουμε ελιάδα σε διοικητικό επίπεδο. Θα πρέπει οι δημόσιες αρχές να συνηθίσουν νέε μεθόδους εργασίας. Μα αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να εξεγερθούμε για αυτό το θέμα. Δεν μπορεί να συνεχίζεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι καλός τρόπος <clears throat> λειτουργίας και σίγουρα αυτό δεν ευνοεί τη δημοκρατική νομιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Σουρμπάν Κρέσπο. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η πραγματικότητα της ανεργίας των νέων για πάνω από 5 εκατομμύρια νέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιδιαίτερα ομοί στην ε, Ισπανία. Οι μισοί νέοι είναι χωρίς δουλειά και απάνω, πάνω από 300.000 νέοι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα μας και ουσιαστικά υπάρχει και μια εκπροσώπησή τους από ένα κόμμα που λέγεται νεότης χωρίς μέλος χωρίς μέλλον. Όλα αυτά οφείλονται στις πολιτικές λιτότητος και δημοσιονομικής προσαρμογής που έχουν ακολουθήσει και το Παρτίδο Ποπουλάρ και το Πεσόε στην Ισπανία. Η τροποποίηση λοιπόν του δημοσιονομικού πλαισίου για να μεταφερθούν κάποιες, ε, κάποια κονδύλια στο 2015 υπέρ της εγγύησης για τους νέους είναι καλό νέο, αλλά είναι ανεπαρκές αυτό το μέτρο. <clears throat> Ας μην αυταπατώμεθα. Για μια ακόμα φορά βρισκόμαστε ενώπιον μιας καλοπιστικής άσκησης. Και πάλι υπάρχει μια πολιτική ενέργεια η οποία δεν εξασφαλίζει την απασχόληση των νέων με ποιότητα και σε απασχόληση με ε, δικαιώματα θα χρειαζόταν μια πολύ μεγαλύτερη ενίσχυση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υποστηρίξουμε κοινωνικές υποδομές, υποδομές που θα είναι χρήσιμες και υποδομές και ενέργειες που θα ήταν σημαντικές για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Ο κύριος Τάραντα έχει το λόγο. Ο κύριος Τάραντα. Ευχαριστώ. Όπως και άλλοι ομιλητές, η προσαρμογή του Πολδίπ προβλέπεται ήδη και το Συμβούλιο, ακόμη και το Συμβούλιο δεν δημιουργεί πρόβλημα. Ο προγραμματισμός των σχεδίων είναι κάτι δύσκολο. Υπάρχουν, σημειώνονται πολλά λάθη γιατί τα κράτη φροντίζουν κυρίως να δαπανούν τα περισσότερα δυνατά χρήματα από την Ένωση παρά την ποιότητα. Αυτό, σε αυτό οφείλονται πολλά λάθη. Η Κομισιόν διστάζει να ελέγξει υπερβολικά τα κράτη-μέλη για πολιτικούς λόγους και ε, στηρίζεται, βασίζεται στα συστήματα ελέγχου των ίδιων των χωρών μελών, πράγμα που είναι πολλές φορές ανεπαρκές. Η ποιοτική δαπάνηση προγραμμάτων ε, είναι κάτι το απαραίτητο. Οι καθυστερήσεις λοιπόν στις πληρωμές και η πρόβλεψη ενός νέου προγράμματος κοινού ελέγχου ε, κομισιών κρατών μελών δεν είναι κακή ιδέα. Έτσι θα διασφαλίζεται η σωστότερη δαπάνηση και απορρόφηση. Φοβάμαι όμως ότι η αναβολή της χρήσης ορισμένων προβλέψεων θα αυξήσει ακόμα περισσότερο την πίεση και τα προβλήματα για τις πληρωμές και το Συμβούλιο φυσικά θα αγνοήσει τις όλο και περισσότερες καθυστερούμενες πληρωμές. Η ομάδα των Πρασίνων με τις 50 ψήφους της θα υποστηρίξει φυσικά την προσαρμογή του Πολδίπα και συγχαίρει και αυτή τον εισηγητή. Κύριος Αρ Νότ. Βλέπω εδώ ότι κανείς δεν είναι κατά. Εγώ εξελέγην για να δείξω, να δώσω μία εναλλακτική άποψη και εμείς είμαστε κατά. Μπορεί να γίνει πολύ καλύτερος τρόπος απορρόφησης των χρημάτων από τα κράτη-μέλη αντί να τα στέλνουν στις Βρυξέλλες για να κακοδαπανηθούν. Διότι το Ταμείο Συνοχής είναι περίπου 33% αυτή τη στιγμή του συνολικού προϋπολογισμού. Αυτό σημαίνει ότι φεύγουν χρήματα από τα κράτη-μέλη και δεν παίρνουν τίποτα σε αντάλλαγμα. Ακούμε ότι 20 δισεκατομμύρια προβλέψεων δεν ε, εκτελούνται. Τι σημαίνει αυτό δεν εκτελούνται. Επιστρέφουν αυτά τα χρήματα στους ευρωπαϊκούς λαούς που τα έδωσαν όσες φορές κύριε Πρόεδρε. Δεν πιστεύουν όλοι ότι η απάντηση σε όλα τα προβλήματα πρέπει να είναι περισσότερη Ευρώπη. Υπάρχει μπλε κάρτα, την δέχεστε. Ορίστε κύριε μου, έχετε το λόγο. Ναι να σας πω για την μπλε κάρτα. Πρόσοχη, γιατί όλα αυτά είναι κατά της πολιτικής συνοχής, όλα αυτά δεν είναι ε, χρήσιμα, λέτε. όμως ξέρετε ότι δεν χρειάζονται αυτά σε κάποιες χώρες για την πολιτική συνοχή, εκεί που γίνονται περισσότερες ε, επενδύσεις, οπότε και έτσι έχουμε ε, βοήθεια στις χώρες εκείνες να ξεπεράσουν την χρηματοπιστωτική κρίση. Το ξέρετε αυτό. Για μένα είναι πάρα πολύ απλό κύριε. Και για το Ηνωμένο Βασίλειο και για άλλα κράτη-μέλη. Στέλνουμε λεφτά στι Βρυξέλλε. Οι Βρυξέλλε τα στέλνουν πίσω. Θα μπορούσαμε το ίδιο αποτέλεσμα να το πετύχουμε. Ακόμα και καλύτερα να τα πάμε. Εάν χρηματοδοτούσαμε κατευθείαν τα σχέδια, προγράμματα, έργα κατευθείαν στα κράτη-μέλη και έτσι να ξέρουν οι κυβερνήσει τι γίνεται. Για μένα είναι πάρα πολύ απλό το θέμα. Ο κύριος Μάρουσικ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, πολλές φορές στην Επιτροπή Προϋπολογισμών τα έχουμε συζητήσει. Τι θα γίνει με αυτή τη μεταφορά των κονδυλίων. Και πολλές φορές το θεωρούμε ένα απλό τεχνοκρατικό θέμα. Όμως, δεν είναι καθόλου τεχνοκρατικό και τεχνικό το θέμα, Πρόεδρε. Είναι κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό και σημαντικό. Γιατί το παρεξηγούμε ότι ο προπολογισμό της Ένωσης είναι κάτι σαν δάνειο προς τα κράτη-μέλη. Προσοχή, γιατί το κόστος είναι πολύ υψηλό. Το να μην χρησιμοποιηθούν κάποια κονδύλια. Οπότε εκεί γίνεται υπέρβαση, έτσι, των ορίων και αποθεματικών. Άρα θα πρέπει να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια. προσοχή επομένως να κάνουμε να προσέξουμε για να είναι καλύτερη η Ευρώπη δημοσιονομικά. Ο κύριος Σντεχόφσκι. Κύριε Επιτροπέ, κύριε και κύριοι. Αυτή η έκθεση δεν είναι μονάχα αφεαυτής σημαντική ω μια τεχνική προσαρμογή για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Είναι και ένα πάρα πολύ σημαντικό πολιτικό μήνυμα. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι πολίτες παρακολουθούν τις ενέργειές μας. Παρακολουθούν τον τρόπο με τον οποίο εμεί αντιδρούμε στις απειλές ενώπιον παραγωγός χάρη στις απειλές εσωτερικής ασφάλειας. Χαίρομαι πάρα πολύ κυρία Επίτροπε που ήλθατε ενώπιον της Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αυτή την πρόταση και με τον τρόπο αυτό συνεχίζεται την επικοινωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο σε πολύ θετικό επίπεδο. Θα να τονίσω ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε την σωστή χρηματοδότηση του Ταμείου για το άσυλο και την μετανάστευση αλλά και για την εσωτερική ε, ασφάλεια που απειλείται από τις ε, μεταναστευτικές αυτές τις ροές. Δεν πρέπει λοιπόν τα κονδύλια αυτά να χαθούν από τα διαφορετικά ταμεία. Θα πρέπει να τεθούν σε κατά προτεραιότητα στους τομείς όπου υπάρχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Πρέπει να υπάρχουν αυτές οι ενέργειες με την κατάλληλη χρηματοδότηση. Και επαναρχόμαι σε αυτό το οποίο είπε και ο κύριος Ντέπρε. Θα πρέπει να εγκριθεί και από το Κοινοβούλιο και από το, από το Συμβούλιο είμαστε ενώπιον μιας κατάστασης η οποία επανέρχεται συνέχεια, λέει ο κύριος Ντενανότ. Όπως είπε και η κυρία Τόμα, θα μπορούσαμε να έχουμε μια καλύτερη λειτουργία για την χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής. Θέλω να υπογραμμίσω την ανάγκη να έχουμε καλύτερη επικοινωνία προς τους πολίτες μας και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες πολύ σπάνια είναι πραγματικά πληροφορημένες για τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο έδαφος τους. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την δυνατότητα μόχλευσης με την χρήση αυτών των πόρων για επενδύσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Κάνω και μία έκκληση για μια καλύτερη και μεγαλύτερη απλοποίηση των διαδικασιών και μεγαλύτερη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών που θα επιτρέψει να υπάρξει μεγαλύτερη ευκαμψία και μεγαλύτερη αξιοπιστία ώστε να μπορούν να προσφεύγουν περισσότερο οι τοπικοί και περιφερειακοί παράγοντες στα διαρθρωτικά ταμεία. Είναι απαραίτητο να τα κάνουμε πιο προσπελάσιμα τα διορθωτικά ταμεία από ό,τι είναι σήμερα, γιατί βλέπουμε όλοι μας ότι υπάρχουν κονδύλια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται. Ενώ θα έπρεπε να είναι οι επιταχυντές των διαδικασιών πλήττονται αυτή τη στιγμή από τη βραδιπορία των διοικητικών αρχών. Ο κύριος Αρτουή. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής και συνάδελφοι, η τροποποίηση του κανονισμού για το πολιτέσμο και πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 βεβαίως και θα πρέπει να επιψηφιστεί. Όμως, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να ε, αναδείξουμε το πόσο έχει γίνει δύσκολη αυτή η διαδικασία και βαριά. Γιατί χτύπησε το καμπανί του κινδύνου όσον αφορά αυτή, αυτό το, το, το, το χρόνιο ε, πρόβλημα. Κάτι το οποίο ε, δεν βοηθάει την ανάκαμψη και μας κρατάει στην ε, υποαπασχόληση γιατί έχουμε αυτά τα 21 δις γιατί έτσι δεν μπορέσαμε να εγκρίνουμε τα προγράμματα οπότε θα πρέπει να υπάρχει διακυβέρνηση θα πρέπει να υπάρχει πολιτική διακυβέρνηση και θα πρέπει η Ευρώπη να μην γίνει ένα τέρας γραφειοκρατικό και τεχνοκρατικό και εγώ λοιπόν κρούω τον κύριο του κινδύνου, τόσο ώστε να απλουστευτούν διαδικασίε αλλά και κείμενε διατάξει. Και κυρία Αντιπρόεδρε, μα αναφέρατε την ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και γι' αυτό θα ήθελα ε, σε αυτέ τι προτάσει σα να καλύψετε και κάποιες ε, προσαρμογές όσον αφορά τις πιστώσεις υποχρεώσεων και πληρωμών ούτω ώστε να δούμε να μην ξαναγίνει αυτού του είδου. Ε, η περικοπή των ε, κονδυλίων για το ορίζον 2020 και για άλλα προγράμματα να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο στο μέλλον. Η κυρία ή ο κύριος Τζάνι, ο κύριος Τζάνι. Πρόεδρε, σίγουρα σήμερα μπορούμε να διορθώσουμε μια κατάσταση ε, γιατί θα πρέπει ομένως πάνω από το 1 τρίτο των κονδυλίων να το μεταφέρουμε για αυτά τα προγράμματα. Γιατί είχαμε μεγάλη καθυστέρηση όσον αφορά την έγκριση αυτών των του 2014 και αυτό την έγκριση αυτών των προγραμμάτων. Επομένω και η Ευρώπη ε, έχει αυτά τα προβλήματα, αυτά που θεωρούμε ότι υπάρχουν μόνο στην Ιταλία. Πρόκειται για κάποιε καθυστερήσει οι οποίε είναι σήμερα σε διάταξη. Οπότε αυτό που θέλω να σα πω είναι ότι και εμεί είμαστε υπέρ του να υπάρχει περισσότερη ε, ευελιξία στο πολιτέ δημοσιογραφικό πλαίσιο και αυτό θα μας βοηθήσει σε πολλές ε, περιπτώσεις να κάνουμε μια τέτοια αναθεώρηση των ε, δημοσιών προοπτικών και επίσης θα πρέπει να μπορέσουμε να κατευθύνουμε τα κονδύλια εκεί που πραγματικά μπορούν να δημιουργήσουν ανάπτυξη ε, και απασχόληση κλπ. Οπότε θα πρέπει να γίνει αυτή η μεταφορά των κονδυλίων και αυτά να χρησιμοποιηθούν επικοδομητικά και να μην διασπαθίζονται ακριβώς όπως έγινε πρόσφατα στην Ιταλία και ε, αυτό να μην φύγει τις περιοχές, τις περιφέρειες που χρειάζονται ακόμη περισσότερο. Κύριε Μοντέλ ο στόχος ήταν να γίνει αυτή η μεταφορά πιστώσεων των 21 δις αυτών των πιστώσεων υποχρεώσεων που δεν χρησιμοποιήθηκαν το 2014, δηλαδή 15% του προπολογισμού του 2014. Πρώτα για μια ε, αναθεώρηση τεχνική, αλλά αυτό σας δείχνει το πόσο σκανδαλώδες είναι η διάθεση των, ε, των ε, των πόρων. Έχουμε επίση αυτά τα, ποσά που δεν έχουν καταβληθεί και αυτό γίνεται γιατί ε, υπάρχει αυτή η γραφειοκρατία. 14,8 δις ήταν όλα αυτά. Ε, μιλάμε για 24 δις και 11 το 2011. Οπότε αυτά όλα θα πρέπει να εκαθαριστούν. Ε, πρόκειται βέβαια για κάποιες περιφέρειες οι οποίες πληρώνουν την ύφη. Οπότε θα πρέπει να δούμε ότι ε, πρόκειται για το πηγάδι πάτο γιατί έτσι χάνονται τα χρήματα και δεν λαμβάνει την υπόψη η εθνική κυριαρχία. Επομένω, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να πάρουν ξανά τα ενία τη κυριαρχία στα χέρια του όσον αφορά τι επενδύσει και αυτού του πόρου. Και να μην ξεχνούμε ότι η Γαλλία δεν ωφελείται και πολύ από αυτό το σύνδεμα Είναι καθαρό εισφορέα των προηγούμενων τη Ένωση. Ε, μιλάμε για 9,4 ε, ε, δις για το 2013. Ο κ. το λέει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, και εγώ χαιρετίζω την προτινόμενη τροποποίηση του πολιετούς ε, δημοσιονομικού πλαισίου και επομένω τον, τον διορθωτικό προπολογισμό 2 για τον οποίο είμαι εισηγητή. Αυτό βέβαια δεν είναι ένα ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο θέμα εδώ στο Κοινοβούλιο. Ο στόχο ήταν τα κρατημένα να μην χάσουν τα κονδύλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία θα αφορούν, <clears throat> αφορούν τα κρατημένα. Ξέρουμε όμω ότι ο κανονισμό του, των διαφορετικών ταμείων και η, η καθυστερημένη έγκριση του πολιετούς προγράμματος οδήγησε σε καθυστερήσεις στα λειτουργικά προγράμματα. Πρέπει να δράσουμε λοιπόν κατεπηγόντως για να αποφύγουμε απώλειες για τα κονδύλια και αυτό είναι απόλυτο ορθό. Για το μέλλον όμως θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, πρέπει να αποφύγουμε <clears throat> όταν θα γίνει η επόμενη ε, η επόμενη έγκριση του πολιτούς πλαισίου να γίνει εγκαίρως και εάν το Κοινοβούλιο κάνει το δικό του έργο θα πρέπει και το Συμβούλιο να πράξει τα απαραίτητα και ζητούμε από την Κομισιόν να είναι έντιμος διαμεσολαβητής ώστε να επιτευχθεί το ταχύτερο δυνατό για να μην υπάρξει και πάλι καθυστέρηση στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Ιδίω σε ένα πλαίσιο οικονομικής κρίσης και σπάνιδος επενδύσεων η έγκαιρη έγκριση των προγραμμάτων και των σχεδίων είναι απαραίτητη για την υλοποίηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για τις επενδύσεις και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρειαζόμαστε και την ανάπτυξη και τι εργασίας περισσότερο από ποτέ. Φυσικά δεν φταίνε μονάχα οι θέσμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη κατάφεραν να εγκρίνουν όλα τα λειτουργικά του προγράμματα και έδειξαν τον δρόμο σε άλλες χώρες όπως η δική μου χώρα η Ρουμανία που υπολείπονται σημαντικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν και προς όφελος των τελικών δικαιούχων να γίνει η έγκριση των λειτουργικών προγραμμάτων ώστε τα ευρωπαϊκά κονδύλια να φτάσουν το λαό της Ευρώπης. Ένα τελευταίο ζήτημα το οποίο θέλω να σας υπενθυμίσω είναι το θέμα των ε, των πιστώσεων υποχρεώσεων για το δεύτερο μισό του δημοσιονομικού πλαισίου και εκεί θα πρέπει η Κομισιόν να κάνει ένα απαραίτητη μέρημνα ώστε να μην χαθούν αυτά τα κονδύλια. Μούντι, η κυρία Μούντι, μαζί με τους άλλους συναδέλφους και εγώ ελπίζω διακαώς ότι θα εγκριθεί αυτό το, αυτή η πρόταση. Τα λειτουργικά αυτά προγράμματα αφορούν τους πραγματικούς, τους απλούς ανθρώπους. Το ξέρουμε πολύ καλά. Στη δική μου περιφέρεια έχω μια κομιτεία η οποία θα πρέπει να λάβει περίπου μισό εκατομμύριο λίρες από το Ταμείο Συνοχής λόγω της αποτυχίας όμως της Βρετανικής κυβέρνησης να ξεκινήσει τα λειτουργικά προγράμματα υπάρχει κίνδυνος <clears throat> να χαθούν τα κονδύλια αυτά και βλέπουμε άτομα τα οποία χάνουν τη θέση εργασίας τους λόγω αυτής της αποτυχίας της Βρετανικής κυβέρνησης να δράσει. Δεν μιλάμε λοιπόν για στατιστικά στοιχεία, μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Υπάρχει όμως και ένα ερώτημα το οποίο εγώ θα ήθελα να θέσω γιατί κάθε πρόγραμμα έχει και μια καταληκτική ημερομηνία, όπως και η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Οποιαδήποτε λοιπόν καθυστέρηση για τα λειτουργικά αυτά προγράμματα μπορεί να σημαίνει ότι θα υπάρχει πολύ περιορισμένο χρονικό παράθυρο για την δαπάνη αυτών των κονδυλίων. Αναρωτιέμαι αν θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε να υπάρχει και ευκαμψία, όχι μόνο τη σύναψη υποχρεώσεων, αλλά και για το χρόνο δαπάνη των κονδυλίων που πρέπει να δαπανηθούν και σωστά για αυτά τα προγράμματα. Η κυρία Πάου Νόβα. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία ε, Γιώργεβα και ε, τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Η μεταρρύθμιση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου για να απευθυνθούν περαιτέρω καθυστέρησης είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Η συζήτησή μας αντανακλά το γεγονός ότι υπάρχει μια ευρεία συνέντευξη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με το θέμα αυτό. Η μεταφορά των πιστώσεων αυτών υποχρεώσεων είναι πάρα πολύ σημαντική για την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού και συνδέεται με τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει να οικοδομήσει μια πιο ευμαρή και ανταγωνιστική οικονομία. Η συμφωνία λοιπόν για το πολιετές πλαίσιο 2014 με 2020 έγινε καθυστερημένα και αυτό είχε επιπτώσεις σε επίπεδο καθυστέρησης των λειτουργικών προγραμμάτων που έχουν φυσικά πολύ σημαντικό αντίκτυπο στις οικονομίες των κρατών μελών και κινδυνεύουν να προκύψουν σημαντικές απώλειες. Εμείς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τους ευρωπαϊκούς πόρους ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη ε, υποστήριξη. Πρέπει όλοι να λάβουν υπόψη το τι μπορεί να τους δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό συμφωνώ με την κυρία Γιώργεβα όταν λέει ότι η Κομισιόν θα πρέπει να συνεργαστεί περισσότερο με τα κράτη-μέλη και τι περιφέρειες ώστε να υπάρξει η σωστή αντιμετώπιση των κονδυλίων αυτών. Τα κράτη-μέλη αυτά λοιπόν δεν μπορούν να καθυστέρησουν περισσότερο, χρειάζονται τη βοήθειά μας για την οικονομική του ανάπτυξη. και δεν συζητούμε τώρα για μια καθυστέρηση των θεσμικών οργάνων. Μιλάμε τώρα για το τι έγινε από πλευρά ε, εθνική, από πλευρά περιφερειακή, τι θα γίνει με σαν προγραμματισμό στο μέλλον. Κυρίω όσον αφορά τα δηλωτικά ταμεία και όσον αφορά την πολιτική τη συνοχή. Επομένω, αυτό που θέλουμε να δούμε τώρα είναι πώ θα υπάρχει ποιότητα όσον αφορά τι ε, πιστώσει, όσον αφορά τα, τα κονδύλια ε, και τι θα γίνει με τι πιστώσει των πληρωμών αλλά και των υποχρεώσεων. Οπότε θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα να επιταχύνει του ρυθμού όσον αφορά αυτά τα τρία μέτωπα. Πρώτα-πρώτα να είναι πιο ε, γρήγορη η έγκριση όλων των προγραμμάτων περιφερειακών και εθνικών. Και επίση θα πρέπει να μην συγκεντρώνονται τα κονδύλια σε ένα συγκεκριμένο έτος γιατί αυτό ε, κινδυνεύει στο να χαθούν κάποια κονδύλια όταν φτάσουμε στην καταληκτική ημερομηνία του 2018 Επίσης χρειάζεται περισσότερη πρωτοβουλία, ούτω ώστε να μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη εμπλοκή των εθνικών υπηρεσιών ερχών σε όλα αυτά. Και έτσι να υπάρξει και αλλαγή νομοθετική για καλύτερο προγραμματισμό και απορρόφηση των κονδυλίων. Σήμερα, Πρόεδρε, ψηφίζουμε αυτήν την τεχνική προσαρμογή και αφορά αυτό, αυτό βέβαια και κάποιες πολιτικές επιλογές. Θα έπρεπε το, το Συμβούλιο να είναι πιο τολμηρό, ούτως ώστε να μπορέσει να, να, να, να αλλάξει το πολιτές πλαίσιο πιο σύντομα. Και έτσι θα, έπρεπε να μην υπάρχουν αυτά τα 21 δις τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν. Και έχουμε τη μεταφορά από το 14 στο 15. Αυτό είναι λογικό. Όμως πολλές φορές δεν επαρκεί η κοινή λογική. Θα πρέπει κάτι να κάνουμε γιατί το πολιετές πλαίσιο θα πρέπει να είναι η βάση επί της οποίας να στηρίζονται όλες οι ευρωπαϊκές πολιτικές. Πριν από μερικές μέρες στην Ιταλία έπεσε ένας πυλώνας, έπεσε ένα στήριγμα γέφυρας. Ο, δεν θα αντικατασταθεί η κολόνα αυτή, θα αντικατασταθεί όλη η γέφυρα για να είναι ασφαλές δηλαδή. Οπότε θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο μετά από αυτή την θητεία θα πρέπει να κάνει μια μετεκλογική αναθεώρηση του πολιτού νομοθετικού πλαισίου. Θα πρέπει αυτό να γίνει ταχαίως και θα πρέπει να γίνει εις βάθος. Ακριβώς όπως έγινε και στην Ιταλία τα παρντέλ. Συνάδελφοι, βρισκόμαστε ενώπιον πολύ σημαντικής πρότασης. Θα πρέπει να αναθεωρήσουμε το νομοθετικό πλαίσιο. Θα πρέπει να διακρίνονται από προβληψιμότητα, από κάποια εφταξία τα κοινωτικά προγράμματα. Μιλάμε για αυτά τα 21 δις του 2014. Θα πρέπει όλοι οι δικαιούχοι τελικά να ωφεληθούν με από αυτήν την τροποποίηση και να δούμε τι θα γίνει με αυτά τα προγράμματα που δεν χρηματοδοτήθηκαν. Όλα αυτά που είναι για την απασχόληση των νέων, για την αντιμετωπιστικότητα της Ευρώπης, αλλά κυρίως τα προγράμματα τα οποία αποσκοπούν σε κοινωνική συνοχή, αλληλεγγύη, ε, για αυτή την περίοδο προβλέπει μέχρι το 18. Οπότε θα πρέπει να δούμε και τι ποσά θα διατεθούν αλλά κυρίως και τι θα γίνει ούτω ώστε να καλυφθούν οι στόχοι που θέλουμε δηλαδή οι μη προνομιούχοι και έτσι να έχουμε μια κοινωνική Ευρώπη πυρήνσκη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η μεταρρύθμιση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου είναι απαραίτητη γιατί υπήρξαν τρεις πολύ σημαντικές τροποποίησεις για την τροποποίηση του πολιτούς πλαισίου, για την έκδοση των κανονισμών για τα Ευρωπαϊκά Διαφορετικά Ταμεία και για την έγκριση των λειτουργικών προγραμμάτων. Επομένως λοιπόν, το 2015 τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δεσμεύσουν τα ποσά τα οποία προβλεπόταν να έχουν δεσμευτεί για το 2014 και 2015 και εξάλλου το 2015 είναι ο τελευταίος χρόνος για την απορρόφηση κονδυλίων από, από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Αυτό σημαίνει μεγάλη πίεση στις αρμόδιες αρχές να σεβαστούν τις ε, ανάγκες για σωστή δέσμευση των κονδυλίων. Μπορεί να υπάρξει λοιπόν και σημαντική αύξηση στον αριθμό των παραβιάσεων για τις οποίες μπορούν να καταγγελθούν τα κράτη-μέλη. Η πραγματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ξεκινήσει με μια πρόνοια να υπάρχει επαρκής χρόνος για την σωστή προετοιμασία και εφαρμογή των κανόνων του προϋπολογισμού. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βόν έχει το λόγο. Πρόεδρε, ε, θέλω να συγχαρώ τους συνεισηγητές γιατί τόνισαν ότι στο τέλος του περσινού έτους μόνο λίγα λειτουργικά προγράμματα είχαν εγκριθεί και είχαμε πει από πέρυσι, από τον Νοέμβριο ότι υπάρχουν καθυστερήσεις και δυστυχώς η Βρετανική κυβέρνηση έδειξε ότι τα λειτουργικά προγράμματα εκεί δεν έχουν καν εγκριθεί ακόμα και αυτό έχει επιπτώσεις για όσους θέλουν να υποβάλουν νέα προγράμματα αλλά και για όσους ενδιαφέρονται για υπάρχοντα που θέλουν να συνεχιστούν. Όλοι όσοι εργάζονται σε αυτά τα σχέδια και όσοι υποφελούνται από αυτά ζημιώνονται βέβαια. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό στο κοινοβούλιο μας σήμερα να δεχτούμε τις αλλαγές, τις μεταφορές των χρημάτων για να αρχίσει η χρηματοδότηση των σχεδίων σε ολόκληρη την Ευρώπη και παρακαλώ την Κομισιόν να πιέσει τα κράτη-μέλη και... Αλλά και αυτό εκείνα να δεχτούν την αλλαγή. Ευχαριστώ. Κύριε Σάντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς θεωρούμε ότι ε, είναι προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη να εφαρμοστούν αυτές οι επενδύσεις είναι δε σκάνδαλο οι καθυστερήσει 21 δισεκατομμύρια από τα διαρθρωτικά ταμεία, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Μετανάστευσης κτλ. Η διαχείρισή τους έγινε κυρίως από τις κυβερνήσεις. Αν γινόταν μάλλον η διαχείρισή τους από τις κυβερνήσεις, ο ρυθμός απορρόφησης μάλλον θα ήταν μεγαλύτερος, υψηλότερο. Τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα πολύ συχνά καθυστερούν λόγω κακής διαχείρισης. Φυσικά το πρόβλημα αυτό το έχουμε από την αρχή της Ένωσης. Μετά όμως το τελευταίο έτος της κρίσης πρέπει επιτέλους να αντιμετωπιστεί η πρόκληση αυτή η εντύπωσή μας είναι ότι οι κρατικοί κανόνες τελικά αντιτίθενται στη σωστή εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων που είναι πολύ υψηλού κόστους και πολύ χαμηλής αποδοτικότητας. Ευχαριστώ. Λιμπεράσκι. Ο κύριος Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω κάπως ανάμεικτα αισθήματα αυτή τη στιγμή σε σχέση με το θέμα αυτό. Από τη μία πλευρά εγώ είμαι υπέρ τα χρήματα αυτά να μην χαθούν, αλλά όλα αυτά γίνονται στο 12 παρα 5 την τελευταία στιγμή πριν από την 1η Μαΐου. Και φυσικά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί αυτή η κατάσταση. Θα πρέπει να καταλάβουμε γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα. Μήπως η αλλαγή της Κομισιόν, η ανανέωση της Κομισιόν έχει συμβάλει. Βέβαια, είναι γεγονός ότι η Κομισιόν έχει ανανεωθεί και αυτό οδήγησε σε κάποιες καθυστερήσεις εξάλλου. Έχουμε και τα καθημέλη τα οποία επέχουν κάποια ευθύνη. Μήπως τα καθημέλη έχουν αυτή τη στιγμή τεράστια επιβάρυνση όταν πρέπει να τελειώσουν και τα προηγούμενα προγράμματα μέχρι το 2013. έχουμε θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ανάλυση για τα θέματα αυτά. Και ένα περαιτέρω ερώτημα στην κυρία Επίτροπο μετά από τα πολλά χρόνια εμπειρίας που έχετε μπορείτε να μας προτείνετε μια απλοποίηση των κανόνων. κύριος Ζουρίνιου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Γίνεται μια ε, μεταφορά ποσών για το 2015 που δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν το 2014. Είναι μια θετική πρόταση η οποία πρέπει να εγκριθεί και ιδίως γιατί συνοδεύεται από μια δήλωση καλή θέληση από την Κομισιόν να μπορέσει να υπάρξει και μεγαλύτερη εμπλοκή των τοπικών και περιφερειακών αρχών για την ε, χρησιμοποίηση αυτών των κονδυλίων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης. Αλλά δεν πρέπει εμείς να επαναπαυόμεθα σε σχέση με το προπατορικό αμάτημα που οδήγησε σε αυτή την κατάσταση τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζετε ότι έχουμε πολλά προβλήματα συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτούν πολύ μεγάλη περαιτέρω επένδυση και είναι απαραίτητο να μην υπάρχει καμία ευκαμψία και η γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπλοκάρει αυτές τις επενδύσεις. Στην Πορτογαλία 16 μήνες μετά από την έγκριση του δημοσιονομικού πλαισίου μόνο τώρα ξεκινούν κάποιοι δημόσιοι διαγωνισμοί και ξεκινούν κάποια προγράμματα. Ελπίζω λοιπόν ότι η έγκριση της σημερινής πρότασης θα επιτρέψει να έχουμε καλύτερη εφαρμογή των δημοσιονομικών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς καθυστέρηση. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στην διαδικασία Catch the Eye με τον κύριο Πεντήρ. Την κυρία Πεντήρ, συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να χαιρετήσω και να καλωσορίσω την πρόταση της Κομισιόν να, ότι θα χρησιμοποιήσει την δήλωση μάλλον της Κομισιόν να χρησιμοποιήσει όλα τα μέτρα για να γίνει κατάλληλη προσαρμογή των δημοσιονομικών των λειτουργικών προγραμμάτων μετά την τροποποίηση του δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020. Τα κονδύλια λοιπόν αυτά τα οποία θα μεταφερθούν στο 2015 για την επίτευξη της εδαφικής συνοχής και της υποστήριξης των φυσικών πόρων θα πρέπει να καταβληθούν για αυτόν τον στόχο. Ελπίζω να μην υπάρξει κάποια τροποποίηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και χρησιμοποίηση αυτών των κονδυλίων σε άλλους χώρους. Όλα αυτά είναι πολύ θετικά για την αγροτική ανάπτυξη, γιατί πολλές χώρες δεν έχουν ακόμα εγκρίνει τα προγράμματά της αγροτικής ανάπτυξης και δεν μπορούν επομένως να χρησιμοποιήσουν τα ποσά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα θέματα λοιπόν της αγροτικής ανάπτυξης και η επιβίωση των πολιτών μας στα χωριά και την Ήπεθρο εξαρτώνται από όλα αυτά. Εμείς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την απασχόληση των ανθρώπων αυτών, τη δυνατότητα να ασκούν τουριστικές δραστηριότητες και να έχουν έτσι κάποιο δίκαιο εισόδημα. Κύριε Καπούτο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου το οποίο δημιουργεί ένα πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο το 2014-2020 έχει εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα αυτό το οποίο προτείνεται τώρα για να συμπληρωθεί αυτό το ε, δημοσιονομικό πλαίσιο ώστε να μην προκύψουν αντικές συνέπειες για τις περιφέρειες και του τελικού δικαιούχου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα βοηθήσει μια πιο ισχυρή πολιτική επενδύσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι απαραίτητο όλα αυτά τα κονδύλια να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά και με μεγάλη ταχύτητα για να δημιουργήσουν ανάπτυξη και απασχόληση που είναι στόχοι που πρέπει να βρισκόνται στην κορυφή των προτεραιοτήτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση του δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 θα πρέπει να εξασφαλίσει την ε, ε λειτουργία των προγραμμάτων που θα έπρεπε να είχαν εκκινήσει νωρίτερα. Είχαμε πάρα πολλέ καθυστερήσει και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Θα πρέπει εξ αυτού να είναι σαφέ ότι η Κομισιόν θα πρέπει μαζί με τα κράτη-μέλη να συνεργαστεί με πιο εφάνταστο τρόπο για να βοηθήσει την ταχύτερη λειτουργία των προγραμμάτων και να υπάρξει μια διευκόλυνση των, διαδικασιών ώστε να υπάρξει πλήρη και επωφελή χρησιμοποίηση όλων των πόρων. Ο κύριος Μαριάς. Πρόεδρε, συμφωνώ με την τροποποίηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 γιατί έτσι πάνω από 300 λειτουργικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και τα υπόλοιπα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορέσουν να υλοποιηθούν ενισχύοντας τις περιφέρειες της Ένωσης. Θα στηριχθεί έτσι η ανάπτυξη και θα περιοριστεί η ανεργία στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και ιδίως στην Ελλάδα που έχει φτωχοποιηθεί από το μνημόνιο θα μπορέσουν έτσι να χρηματοδοτηθούν αναπτυξιακά έργα στην ελληνική περιφέρεια από το ταμείο συνοχής. μέσα από το ευρωπαϊκό γεωργικό ταμείο αγροτικής ανάπτυξης μπορούν να ενισχυθούν οι πλημμυροπαθείς αγρότες στα τενάγη των φιλίππων στις σέρες και στον εύρο. από το ταμείο ασύλου και μετανάστευσης θα υπάρξει αρρωγή στην ελλάδα που κινδυνεύει να γίνει νέα λαμπεντούζα λόγω των χιλιάδων προσφύγων που σειραίουν στα νησιά του αιγαίου. τέλος καταγγέλουμε από το βήμα αυτό την εκβιαστική πολιτική της τρόικας που έχει παγώσει την εκτέλεση στην πατρίδα μας των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ευρωπαϊκή ένωση προκειμένου η ελλάδα να υποκύψει στην εκβιαστική πολιτική των δανειστών. ευχαριστώ. Παρά το ότι το θέμα είναι τεχνικό, γιατί πρόκειται για μια νομική αλλαγή, πρόκειται και για μια σοβαρή πολιτική απόφαση. Ποια είναι αυτή η σοβαρή πολιτική απόφαση δε, είναι η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε μια κατάσταση όπου 21 δισεκατομμύρια προβλέψεων που έχουν χορηγηθεί δεν πληρώνονται μήνες και χρόνια διότι όσοι πιστεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές απευθύνονται, υποβάλλουν τέτοια σχέδια και έτσι θα χάσουν την πίστη τους στην Ένωση. Γι' αυτό υποστηρίζω αυτά που είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές και ως άνθρωπος που ασχολήθηκε με 300 τέτοια προγράμματα και σχέδια θα ήθελα να καλέσω την Κομισιόν να απλοποιήσει τις διαδικασίες. Ευχαριστώ. με ικανοποίηση δεχόμαστε αυτό το μηχανισμό ευκαμψίας που θα επιτρέψει οι πόροι που δεν χρησιμοποιήθηκαν το 2014 να μεταφερθούν στα επόμενα χρόνια. Αυτό ήταν κάτι το οποίο μπορούσε κανείς να προβλέψει αν λάβει υπόψη την καθυστέρηση των διαδικασιών στο νέο πλαίσιο. Σε επίπεδο αγροτικής πολιτικής και ιδίω σε επίπεδο αιτήσεων για τις επιδοτήσεις υπήρξαν ανάγκες, υπήρχαν ανάγκες μεγαλύτερης ευκαμπτοποίησης από την Κομισιόν. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε σε αυτή τη συζήτηση ότι το πολιτές πλαίσιο ενώ δηλώνει ότι είναι υπέρ μιας κοινωνικής Ευρώπης δεν δίνει τα απαραίτητα κονδύλια να ξεπεραστούν οι ανισομέρειες και οι ανισότητες σε μια εποχή που η Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει μια μεγάλη κρίση. Επίσης δεν μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί δεν χρησιμοποιούν χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση πόρους σε σημαντικό επίπεδο για να εξασφαλίσει την ε, ε, αξιοπιστία της και ζητά τα κράτη-μέλη να κάνουν κάτι το οποίο δεν μπορούν λόγω της λιτότητας να φράξουν. Ο κύριος Σόλτες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Πιστεύω ότι από τη σημερινή συζήτηση γίνεται σαφές ότι η τροποποίηση αυτή του δημοσιονομικού πλαισίου θα γίνει δεκτή και η πρόταση της Κομισιόν θα πρέπει να υποστηριχθεί ώστε τα κονδύλια αυτά να μπορέσουν να μεταφερθούν στο έτος 2015. Υπάρχουν όμως και ελοχεύοντες κίνδυνοι. Κίνδυνοι να είναι μεγαλύτερο το ποσοστό σφαλμάτων και το ελεκτικό συνέδριο έχει ήδη επισημάνει ότι υπήρξαν πολλά προβλήματα στην εφαρμογή των κονδύλιων και δεν έχει επιληθεί το σύνολο των προβλημάτων αυτών. Αίτιο είναι η πολυπλοκότητα των διαδικασιών που οδηγεί πολλέ φορέ σε παραλήψει. Αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση λοιπόν για την Κομισιόν η οποία θα πρέπει να εκπληρώσει αυτό το οποίο έχει υποσχεθεί. Δηλαδή να απλοποιήσει τις διαδικασίες. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε μονάχα τα θέματα της γραφειοκρατίας. Θα πρέπει να σταθούμε στην ουσία των σχεδίων και να καταλάβουμε ποιοι είναι οι λόγοι των αποτυχιών και να τους θεραπεύσουμε. Παρόλ. Euh, euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε θα σας πω ότι συμφωνώ να υπάρξει αυτός ο τροποποιητικός κανονισμός για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020. Θα έχει θετικά αποτελέσματα αυτή η αλλαγή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη και την ανάκαμψη στην Ευρώπη. Η νέα πολιτική συνοχή θα στηρίξει τις καινοτόμες επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βιώσιμη απασχόληση, τις ε, δεξιότητες, θα υπορμήσει τη φτώχεια, θα βοηθήσει τα ευρυζωνικά στις περιφέρειες, το περιβάλλον, ενεργειακή, τη χρήση της ενέργειας και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις μεταφορές και τις διασυνδέσεις θα βοηθήσει την δημόσια διοίκηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια έγκαιρα, όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά για ανάπτυξη και απασχόληση. Ελπίζω να εγκριθούν συντόμως ε, οι και τα προγράμματα που δεν έχουν εγκριθεί και με ρεαλισμό να υπάρξει αύξηση της προοικοδότησης. Σας ευχαριστώ. Γκραπίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους εισηγητές αλλά και την αρμόδια Επιτροπή του Κοινοβουλίου. Χρειαζόταν αυτή η αναθεώρηση. Είναι πολύ σημαντικό σήμερα να εγκρίνουμε αυτή την πρόταση. Γνωρίζουμε τα προβλήματα, αυτά που αντιμετωπίσαμε το 2007-2013. Υπάρχει αυξημένο κόστος, δαπάνες, ε, υπάρχει πολλή γραφειοκρατία θα πρέπει να απλουστευτούν οι σχετικές διαδικασίες αλλιώς και στο μέλλον θα έχουμε τα ίδια προβλήματα. Θα πρέπει το Ταμείο Επενδύσεων να βοηθήσει και να γεφυρθούν τα χάσματα μεταξύ των περιφερειών. Και ε, έχουμε και τις προτάσεις Juncker που θα βοηθήσουν οπότε θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και κάποια γεωγραφικά κριτήρια, θα πρέπει να λάβετε υπόψη τις διαφορές για την επιλογή των εμπειρογνωμόνων ούτω ώστε να χρησιμοποιηθούν αυτά τα κονδύλια και να γεφυρωθεί το χάσμα ε, μεταξύ των περιφερειών. Θα πρέπει να υπάρξει εγγραφτικός έλεγχος και ελπίζουμε ότι, ότι στο μέλλον τα πράγματα θα είναι καλύτερα από ότι τώρα. Κύριε Γεωργίευα, έχετε το λόγο, λέει ο πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους όσους έλαβαν το λόγο και εκφράστηκαν υπέρ αυτής της πρότασης. Θα σα αναφέρω τέσσερα ζητήματα σε σχέση με τις παρατηρήσεις, τις ερωτήσεις που μας ε, απίθυνα οι βουλευτές πρώτα-πρώτα όσον αφορά τις επιπτώσεις για τις πληρωμές. Όπως βλέπουμε εμείς τα πράγματα, θεωρούμε ότι τα πράγματα είναι πιο διαχειρίσιμα Past payment profile. όσον αφορά το πώς γίνονται πληρωμές στο παρελθόν. Αλλά επίσης έτσι θα βγούμε από αυτό το αδιέξοδο των πληρωμών γιατί συνεργαστήκαμε με καλά αποτελεσμένα τα κρατημέλη και έτσι κάναμε την προβολή των εκταμιεύσεων για πληρωμές και έτσι μπορούμε τώρα να διαρθρώσουμε τις ε, πληρωμές με έναν πιο προσεκτικό τρόπο, πιο προβλέψιμο τρόπο. Επίσης υπήρχε μία ερώτηση που υπευλήθη σε σχέση με τις χώρες που δεν θα μπορέσουν να απορροφήσουν αυτά τα κονδύλια. Έχουμε τον κανόνα νη συν 3. Ισχύει ο κανόνα αυτό, θα εφαρμοστεί. Και αυτό σημαίνει ότι άπαξ και γίνει η ανάληψη των υποχρεώσεων υπάρχει ο αναγκαίος χρόνος ούτως ώστε να εκτελεστούν τα εγκριθέντα προγράμματα. Και ε, κάνω σε αυτό σημαίνει ότι έχουμε τρία χρόνια παραπάνω από όσο κρατάει το, ε, το δημοσιονομικό πλαίσιο. Αρχές ε, επομένου έτους θα γίνουν κάποιες εγκρίσεις άλλε πιο μετά. Τέλο πάντων θα χρησιμοποιηθούν όλα αυτά τα χρήματα. Και επίση σα τονίζω και πάλι ότι αντιλήσαμε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα από αυτή την κρίση ρευστότητα. Και έτσι μάθαμε το πώ μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα τη σχέση υποχρεώσεων και πληρωμών στα πλαίσια του υποπολογισμού. Πέρασε η εποχή των παχαίων αγελάδων. Πρέπει να δουλεύουμε σε σφιχτό διαμηνοσομικό περιβάλλον. Και θα πρέπει επομένω να προσέχουμε και την ποιότητα της ανάλωση των πόρων και όχι μόνο τα κόστα. Οπότε κάτι άλλο το οποίο αφορά την απλούστευση γιατί το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο από εσά. Είπατε ότι πρέπει να έχουμε απλούστερες διατάξεις ούτω ώστε τα προγράμματα να εκτελούνται όπω πρέπει να υπάρχουν λιγότεροι κίνδυνοι, οπότε εμεί θεωρούμε ότι αυτό είναι θέμα υψηλή προτεραιότητα. Παρακαλώ, συνεργαστείτε. Να μην προσθέσουμε νέες διατάξεις για ελέγχου εκεί που δεν χρειάζονται, εκεί που δεν φέρνουν κάποια προσθέμενη αξία. Αλλά θα πρέπει να συνεργαστούμε και με τα κράτη-μέλη. να έχουμε αυτούς τους ελεκτικούς κανόνες ε, υπάρχουν ρήτρες διασφάλισης, υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες. The value for money is this something that should be supported. There were voices saying, let's just... Και όπου χρειάζεται να μπορούμε να προσθέσουμε κάτι μέλη στο κανονιστικό πλαίσιο. Τώρα κάτι άλλο. Θέλω να πούμε κάτι επί τη βάση των ε, στοιχείων και πραγματικών περιστατικών. Οι, οι πόροι ε, της συνοχής αφορούν και τις χώρες δικαιούχους αλλά και όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν αναλύσουμε λοιπόν τα, τα, τα, τους πόρους αυτούς στην προηγούμενη θα δούμε ότι άμεσα επηρέασαν την ανάπτυξη. 2,1% για τη Λετωνία και 8,1% για τη Λιθουανία, για την Πολωνία 1,7% και επομένως ε, έχουμε περισσότερες θέσεις απασχόλησης αλλά αυτό σημαίνει και αγοραστική δύναμη. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο αφορά ε, κάποια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί αναφέρεται ότι έχουμε την πιο αποτελεσματικό, τον πιο αποτελεσματικό μηχανισμό μετατροπής δηλαδή ε, κάποιος περνάει πάρα πολύ εύκολα από το μεσαίο εισόδημα στο υψηλό εισόδημα. Πρόκειται για ένα άλμα, το πιο δύσκολο. Και 12 ώρες το κατάφεραν αυτό. Είναι χώρες που βρήκαν πετρέλαιο, οι μισές, και άλλες μισές είναι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανείς ανταγωνισμό πάρα πολύ αυστηρή. Εμείς πολλές φορές που υπερβάλλουμε όσον αφορά το πόσο δημοκρατικοί είμαστε πάντως θέλουμε ανάπτυξη χωρίς να αυτό να είναι εις βάρος της δημοκρατίας της καταπολέμησης της περιθωριοποίησης της κοινωνικής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φυσικά σεβόμενοι και την αλλαγή του κλίματος. Τώρα όσον αφορά τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση έλαβε υπόψη ότι είπατε που είναι πολύ αξιόλογα. Βεβαίως και θα κάνουμε μια ενδελεχή ανάλυση για το κατά πόσον το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο αντικατοπτρίζει αυτά που πρέπει, την πραγματικότητα και τις προτεραιότητες. Όπου χρειάζεται θα κάνουμε προσαρμογές και βέβαια αυτές οι προτεραιότητες εάν απαιτούν αναθεώρηση, ε, τότε εμείς θα προτείνουμε την κατάλληλη αναθεώρηση και σας τονίζω θα χρησιμοποιήσω το νέο μέσο ευελιξίας για αυτές τις προτεραιότητε και αυτό το συνολικό πλαίσιο για τις υποχρεώσεις. Θα συνεργαστούμε με τον κύριο Αρτουή, την Επιτροπή Προπολισμών, με το Κοινοβούλιο και έτσι τα χρήματα των φιλολογουμένων να πηγαίνουν για το καλό της οικονομίας μας και των Ευρωπαίων. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Τομά, χρησιμοποιήσατε όλο το χρόνο που είναι διαθεσή σα, αλλά τέλος πάντων ξανά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, ευχαριστώ και γνώριση του κυρίου Όλμπριχτ που δεν μπορούσε να παραστεί εδώ τα περισσότερα που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας βρίσκουν σύμφωνος τους περισσότερους εξημών ευχαριστούμε για τις εξηγήσεις σας κυρία Αντιπρόεδρε Πέραν αυτό που είπατε βέβαια και για, τα, για τις πληρωμές, θεωρούμε ότι όλα αυτά είναι καλά μαντάτα. Επομένως δίνουμε ραντεβού για να δούμε πώς θα γίνει αν χρειαστεί η αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου που θα είναι ουσιαστική αναθεώρηση και όχι απλά τεχνική αυτή τη φορά.